μετά το ψήφισμα την πραγματικότητα, τα πραγματικά γεγονότα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μίρσκι. Στο τέλος η κυρία Μπασέσκου. Κύριε, κύριε Πρόεδρε, μια πολύ σημαντική πτυχή της σημερινής συζήτησης ήταν η